ξεκινήσουμε μια ευρεία συζήτηση για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά για την ενσωμάτωση των Ρώμα. Το τον έκλεισε έκλεισε συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Αύριο στις 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 και από τις 3 έως τις 9 θα συνεδριάσουμε πάλι. Ε, έχετε το, την ατζέντα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου